commencer. Voilà. Si vous le voulez bien, on va commencer. Ça fera venir les autres. Ça attirera nos collègues pour cette séance dont l'ordre du jour a quand même beaucoup d'intérêt sur le fond. Καλημέρα σα. Να αρχίσουμε, θα έρθουν και οι άλλοι σιγά σιγά. Το σχέδιο μερίσια διάταξη μα μπορούμε να το εγκρίνουμε αν δεν διαφωνείτε τώρα 18 Ιανουαρίου τα πρακτικά, να τα εγκρίνουμε επίση αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, ε, ε, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει μέχρι το τέλος της ε, πρωινή συνεδρία. μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν ε, στην ημερήσια διάταξή μας. Το πρώτο σημείο της ημερήσια διάταξης ε, αφορά ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό για τους σιδηροδρόμους που είναι το σύστημα διαχείρισης ε, της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, το ERTMS. Ξέρετε ότι είναι ένα σύστημα πάρα πολύ σημαντικό για τη συνοχή, την καλή λειτουργία των σιδηροδρόμων μας. Έχουμε όμως ακόμη πάρα πολύ δρόμο μέχρι να επιτύχουμε το στόχο μας δηλαδή η παρουσία, την παρουσία του συστήματος αυτού ε, με τρόπο διαλειτουργικό ώστε να επιτρέπει και στους επιβάτες αλλά και στα εμπορεύματα μια καλύτερη μεταφορά. Είμαστε λοιπόν πάρα πολύ μακριά παρά το γεγονός ε, ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς ε, κάνουν πολύ θετικές δηλώσεις. Είναι κάτι δύσκολο και οικονομικά και πολιτικά. Είναι εδώ ε, ο κύριος Λάτισλαφ Μπάλκο, τον οποίο ευχαριστώ που είναι εδώ σήμερα μαζί μας ε, είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και είναι εισηγητής για την ειδική έκθεση του ERTMS ε, και ο οποίος θα μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα του πρόσφατου ελέγχου του συνεδρίου. Θα ήθελα να καλωσορίσω και τον κύριο Κέρφιτς ε, από την DG Move της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θα μας παρουσιάσει το έγγραφο εργασίας προσφάτως δημοσίευσε η Επιτροπή σε σχέση με το μέλλον του ERTMS. Κύριε Μπάλκο, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Ε, κυρίες και κύριοι, Κυρία Εισηγήτρια, κύριε Πρόεδρε, η δική μας Επιτροπή 13 του 2017 σε σχέση με το ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης ε, της ε, ε, σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, αν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα, είναι μία ακόμη, ένας, μία ακόμη έκθεση για την επίδοση του συστήματος αυτού και το καλοκαίρι θα παρουσιάσουμε ε, και μία έκθεση για τους σιδηροδρόμους ταχείας, όπως επίσης και μία επισκόπηση του, ε, των μεταφορών και της κινητικότητας. Εγώ θα ήμουν εισηγητή στην προηγούμενη μας έκθεση, 8-2016, για τις μεταφορές εμπορευμάτων. Ε, διαπιστώσαμε ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Σιδηροδρόμων είναι, αποτελείται από διαφορετικά εθνικά συστήματα, τα οποία δεν είναι απολύτως διαλειτουργικά και είχαμε σημειώσει ιδιαίτερος ότι το ERTMS ε, τύχανε πολύ αργής αφορμογής. Η τρέχουσα έκθεσή μας ε, βασίζεται στην έκθεση για τα εμπορεύματα. Ιστορικά οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναπτύξει τις δικές τους τεχνικές προδιαγραφές για τα συστήματα σηματοδότησης των σιδηροδρόμων που δεν είναι διαλειτουργικά. Για να μπορέσουμε να το υπερβούμε αυτό και να δημιουργήσουμε μια ενιαία, έναν ενιαίο χώρο σιδηροδρόμων ε, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπή στα τέλη του 1980 άρχισε να αναπτύσσει το ERTMS με σκοπό να, να, να, αντικαταστήσει τα συστήματα σηματοδότηση στα εθνικά για να μπορέσουν τα τρένα να λειτουργούν ανεμπόδιστα μεταξύ των χωρών και να υπάρχει και ανταγωνιστικότητα η συμβολή από τα διαρθρωτικά ταμεία και τα διευρωπαϊκά ταμεία ήταν 1,2 δις ευρώ στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και 2,7 δις ευρώ στην τρέχουσα περίοδο. Ε, η σωστή ε, λειτουργία προκύπτει από ε, την καλή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των προγραμμάτων και πρέπει να υπάρξει μια πραγματική ανάπτυξη βάσει διαχειριστών υποδομής ε, και φορέων εκμετάλλευσης που θα έχουν στη διάθεσή τους το ERTMS. Έχουμε εξετάσει κατά πόσο το σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και τύχει σωστής διαχείρισης. Ε, η Δανία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, οι κάτω χώρες και η Πολωνία εξετάστηκαν. Ε, καλύπτουμε όλους τους διάδρομους του κεντρικού δικτύου που πρέπει να αναπτυχθεί το ERTMS μέχρι το 2030. Επίσης αναπτύξαμε, επίσης είδαμε τα 26 ε, δείγματα ε, σιδηροδρομικών εταιριών σε όλα τα κράτη-μέλη και θεωρούμε ότι το σύστημα, ότι το ERTMS για την ώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ένα χαμηλό επίπεδο ε, λειτουργίας. Ε, χρειάζεται οι φορείς εκμετάλλευσης να κάνουν ε, επένδυση σε πολύ δαπανηρή υποδομή ε, και δεν υπάρχει ένα επαρκές επιχειρηματικό μοντέλο για όλους τους ε, μόνο ένα μικρό ε, τμήμα της δαπάνης μπορεί να καλύψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο θέτει ένα αμφιβόλο όχι μόνο του στόχους του 2030 για το βασικό δίκτυο και τις επενδύσεις ως τώρα, αλλά επίσης και για την υλοποίηση ενός ενιαίου χώρου ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων και Τη ανταγωνιστικότητα ε, του σιδηροδρόμου σε σχέση με τις οδικές μεταφορές. Πιο συγκεκριμένα, σε σχέση με τον προγραμματισμό του ERTMS, διαπιστώσαμε ότι παρά την στρατηγική πολιτική επιλογή ανάπτυξης ενός ενιαίου συστήματος σηματοδότηση ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπήρξε πλήρης ε, εκτίμηση των αναγκών χρηματοδότηση για το πλήρε δίκτυο το κεντρικό. Οι νομικέ υποχρεώσει που υπήρξαν ε, ε, δεν, υπήρξαν, δεν ήταν πάντοτε ευθυγραμμισμένε με ε, την πολιτική μεταφορών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη, από τα κράτη-μέλη μόνο η Δανία κατάφερε να απομακρύνει το εθνικό τη σύστημα υπέρ του ERTMS. Για τα υπόλοιπα κράτη που εξετάστηκαν είναι απλώ ένα επιπρόσθετο σύστημα στα εθνικά του συστήματα. Το επίπεδο τη ανάπτυξη του συστήματο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι χαμηλό, πρόχειρο και υπάρχουν πολλά κομμάτια τα οποία δεν συνδέονται με τα υπόλοιπα. Το στα τέλη του 2016 μόνο 8% του, των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου ε, λειτουργούσαν ε, εντός του συστήματος ERTMS. Είναι λοιπόν χαμηλή, ε, χαμηλό το ποσοστό ε, ανάπτυξης και εφαρμογής, όμως θεωρούμε ότι υπάρχει καλός συντονισμός. Κάνουμε λοιπόν τι εξή δύο συστάσει. Καταρχά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη πρέπει να αναλύσουν το πλήρε κόστο του ERTMS και τη ανάπτυξή του ανακράτο μέλο. Και δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ζητήσει ε, να υπάρξει μια συμφωνία με, τα κράτη-μέλη για ρεαλιστικού, συντονισμένου και νομικά δεσμευτικού στόχου ε, για τον παροπλισμό των εθνικών του συστημάτων ε, σηματοδότηση. Όσον αφορά την ανάπτυξη για το επιχειρηματικό μοντέλο, είναι ένα ενιαίο σύστημα για πολλούς ε, ε, χειριστές υποδομών και φορείς εκμετάλλευσης με διαφορετικές ανάγκες. Είναι δαπανηρές οι επενδύσεις που χρειάζονται, χωρίς άμεσο αποτέλεσμα, ε, κυρίως για όσους πρέπει να φέρουν το, κόστο, το βάρος του, κυρίου, του μεγαλύτερου κόστους, ανεξαρτήτως του, του γενικού θετικού αποτελέσματος στο μέλλον, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επειδή πρέπει να ολοκληρωθεί το ERTMS και να αντικαταστήσει τα εθνικά συστήματα ε, υπάρχουν προβλήματα συμβατότητα, Για την ώρα δεν υπάρχει μία μονάδα ε, σε όλους τους σιδηροδρόμους που να δίνει τη δυνατότητα λειτουργία του ERTMS σε όλα τα τμήματα ε, του σιδηροδρομικού δικτύου τα κράτη-μέλη επέλεξαν την ανάπτυξη του ERTMS σε διαφορετικά στάδια της ανάπτυξής του και σε, και σε διαφορετικές γραμμές των δικτύων τους. Έχουν εξελιχθεί οι τεχνικές προδιαγραφές για τη διατηλειτουργικότητα πολύ γρήγορα, κάτι το οποίο παρεμποδίζει την συνολική σταθερότητα του συστήματος και έχει ε, ως αποτέλεσμα πολλές αναβαθμίσεις. Θεωρούμε παρόλα αυτά ότι το ERTMS δημιουργεί κάποια ωφέλη για τους ε, χειριστές και τους φορείς εκμετάλλευσης ε, των σιδηροδρομικών δικτύων όσον αφορά την ταχύτητα και την ε, ε, ε χωρητικότητα. Το 2014 έπηξε ένα, πρόγραμμα, ε, ένα νέο πρόγραμμα και, και το 2017 ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης παρά τα οποία ε, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις. Δεν υπάρχει ακόμη ας πούμε, νομικά δεσμευτική προθεσμία για τον παροπλισμό των εθνικών συστημάτων. Επίσης, οι διαδικασίες πιστοποίησης είναι πάρα πολύ χρονοβόρες. Πιστεύουμε όμως ότι ο ενισχυμένο ρόλο ε, του, του Οργανισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση για του Σιδηροδρόμου, που το 2019 θα γίνει το επίσημο σύστημα για τη λειτουργία του ERTMS υπό το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο, είναι ένα βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση. Βάσει αυτών των παρατηρήσεων για την ανάπτυξη του ERTMS, ε, προβαίνουμε στι εξή ακόμη συστάσει. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη πρέπει από κοινού με του εμπλεκόμενου φορεί και ε, τους υπεύθυνους του ERTMS να εξετάσουν τους διάφορους ε, χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για την υποστήριξη των επιχειρηματικών μοντέλων για την ανάπτυξη του ERTMS, ε, να μην περιμένουν επιπρόσθετη βοήθεια από τον Ενωσιακό Προπολογισμό. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ERA πρέπει με την υποστήριξη ε, πρέπει ε, να συνεχίσει να ε, διορθώνει τα σφάλματα που εξακολουθούν να υφίστανται, να μην υπάρχουν πλέον προβλήματα συμβατότητας, αλλά να υπάρχει συμβατότητα για όλα τα, όλες τις γραμμές που έχουν το σύστημα ERTMS. Πρέπει να μπορεί να υπάρχει ένας χάρτης για την ανάπτυξη ενός τυποποιημένου συστήματος για όλα τα τμήματα του δικτύου και να υπάρξει και μια διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμών για να μπορέσει να ε, βελτιωθεί το σύστημα ERTMS. Τρίτον, το Ευρωπαϊκό, το Ευρωπαϊκή, Επιτροπή πρέπει να δει κατά πόσο ο ERA έχει τις, ε, τους απαραίτητους πόρους για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ε, ευθύνες του. Και τέταρτον, τα κράτη-μέλη πρέπει να ευθυγραμμίσουν τα εθνικά προγράμματα ανάπτυξή τους και να αναπτύξουν, να συντονίσουν τις προθεσμίες ανάπτυξης του προγράμματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί και να επιβάλλει την εφαρμογή του νέου συστήματος Ανάπτυξης και να θέσει ορόσημα για τη σωστή παρακολούθηση της πρόοδου. Και τέλος, ως την ε, ως προς τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση του ERTMS υπάρχει ε, και, για τις, ε, και για τις τροχές αλλά και μέσα στις ε, αυτοκινητάμαξες όμως μπορεί να καλύψει ένα μικρό τμήμα του συνολικού ε, κόστους ε, δεν μπορεί πάντοτε να καλύψει τα πάντα εμείς αξιολογήσαμε το μέγεθος των επενδύσεων που μπορεί να χρειάζονται για να υπάρξει ένα λειτουργόν ERTMS ε, σε όλο το κεντρικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και το κόστος είναι περίπου ε, κάτι ανάμεσα σε 73 και 177 δις ευρώ όσον αφορά τον εξοπλισμό ε, στους σιδηροδρόμους θα μπορούσε να φτάσει μέχρι τα 80 δις για το κεντρικό δίκτυο και 190 δις για το συνολικό δίκτυο. Μπορείτε να δείτε την τεράστια διαφορά σε σχέση με την ε, χρηματοδότηση του 1,2 δις ευρώ στο προηγούμενο πρόγραμμα, στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και 2,7 δις στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο το τροχαίο, για το τροχαίο υλικό ε, το κόστος ε, είναι διαφορετικό ε, ανάμεσα μεταξύ των μηχανών που χρειάζεται να αναπροσαρμοστούν με το ERTMS και των νέων μηχανών ε, ένα δις ε, μπορεί ε, να είναι η προσαρμογή του κάθε, της κάθε μηχανής και το μέσο κόστος εξοπλισμού των, της νέας μηχανής είναι περίπου 300.000 ευρώ ή 15% της αξίας της μηχανής δεν χρησιμοποιούνται όλοι, όλη η χρηματοδότηση δεν χρησιμοποιείται για τα project του ERTMS. 50% των διευρωπαϊκών δικτύων και των, της χρηματοδότησής τους αρχικά είχε διατεθεί για το, για το ERTMS, ε, όμως στα κράτη-μέλη ε, που επισκεφθήκαμε το ποσοστό απορρόφησης ήταν 86%. Ελπίζουμε ότι ε, υπάρχει ένας κίνδυνος ε, η, ε, τα, τα, τα κονδύλια του, της, του συνδέοντας την Ευρώπη μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την περίοδο 2014-2020 γιατί τη στιγμή του ελέγχου μας μόνο 50 εκατομμύρια είχαν εκταμιευθεί. Επίσης καταφέραμε Επίσης είδαμε ότι υπάρχει ανεπαρκής στοχοθέτηση ε, ως προς ε, τις ε, μονάδες ε, του κεντρικού δικτύου. Ε, επίσης κάνουμε και το τελευταίο μας σύνολο συστάσεων που είναι το εξής. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να, ε, προσαρμόσει ε, το συνδέοντα στην Ευρώπη για να μπορέσει να μεγιστοποιήσει την απορρόφηση των... Ε, της χρηματοδότησης με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι υποφελής για το ERTMS και δεύτερον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη πρέπει να θέσουν καλύτερους στόχους σε σχέση με την περιορισμένη χρηματοδότηση που υπάρχει για τα project του ERTMS Πρέπει η χρηματοδότηση να αφορά κυρίω διασυνοριακά, αν υπάρχει κατά προτεραιότητα για διασυνοριακά τμήματα ή για του ε, τους διαδρόμους του κεντρικού δικτύου ε, και πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στους φορεί εκμετάλλευση σιδηροδρόμων που συμμετέχουν περισσότερο στο διεθνή, στις Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε να πούμε ότι είναι θετική ανάλυση του ελληνικού συνεδρίου ε, και έχουμε συνεργαστεί αποδοτικά με τον κύριο Μπάλκο και το να τονίσουμε αυτό χρησιμοποιείται παντού στην Ευρώπη για τους αισθητοδρόμους Αυτό ήταν κατόρθωμα γιατί όπως είδατε από την έκθεση να σας πω για το πρόγραμμα δράσης και τα επιμέρους σημεία του. Όμως Άζει σκληρό τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την ε, ε θέσπιση αυτού του τέταρτου ψηφοδρομικού πακέτου. Επομένω, το πιο σωστό τώρα είναι να λειτουργήσει για να μην ξανααλλάξουμε ε, μέθοδο και πολιτική. Και η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού προβληματίστηκε και επομένω έχει γίνει και οικονομική ανάλυση που συνοδεύει αυτές τις ε, επιπτώσεων σε έκθεση όπως το είπε ο κ. Μπάλκο. Το πρώτο ζήτημα είναι για το αν, έχουμε, αν έχουν πιάσει τόπο οι κοινοτικοί πόροι. Όντω, έγιναν σημαντικά βήματα όσον αφορά το ΣΕΦ, το Connecting Europe Facility. Κατά τα λοιπά ε, είμαστε στο μήκο κύματο του ελεγκτικού συνεδρίου όσον αφορά τι προτεραιότητε, όσον αφορά τα σημαντική πρόοδο σε σχέση με την αφετηρία αυτή της πορεία του 2007. Τώρα όσον αφορά το 80 και το 90 είναι σημαντικό να αναγνωρίσει κανείς ότι αυτό το πρόγραμμα δεν το επιβάλαμε στα κράτη-μέλη ούτε όσον αφορά το υψηλό κόστος της ανάπτυξης. Εδώ έχει κάποιες ε, αποκρισταλωμένες απόψεις το ελεγκτικό συνέδριο πώς το ERTMS θα αναπτυχθεί στο μέλλον βεβαίως και πρόκειται για μια πρόκληση αλλά εμείς χρειάζονται ε, αντικαταστάσεις χρειάζονται αντικατάσταση κάποια κομμάτια του συστήματος, ούτω ώστε να υπάρχει ασφαλής κυκλοφορία των σιδηροδρόμων. Το τι γίνεται όσον αφορά την ε, μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο. Πρόκειται ακριβώ για αυτέ τι αλλαγέ που έπρεπε να γίνουν για να προχωρήσουμε. Όπω τα λέει και η έκθεση, πάμε τώρα στην τρίτη διαφάνεια. Εδώ έχω εφαρμογή τη υλοποίηση. Εδώ έχουμε τις ε, συγκεκριμένες ε, ε, συνταγές οι οποίες είναι συμπεφωνημένες με την βιομηχανία. Άρα βλέπουμε ότι η αρχή των σειροδρόμων θα έχει τώρα αυξημένες αρμοδιότητες. Να δούμε πώς θα υπάρχει κάποια ομοιογενής εφαρμογή του ERT και έχουμε ορόσημο το 2023 για τις ε, γραμμές που θα είναι λειτουργικές μέχρι τότε. Πάμε τώρα στην τέταρτη διαφάνεια. Εδώ έχουμε κάποια τμήματα. Παρουσιάζει ενδιαφέρον αυτό για την ε, βιομηχανία, για τους εμπλεκομένους και όπου υπάρχουν ε, δυσκολίες για κάποιους εμπλεκομένους, τότε θα πρέπει η Ένωση με χρηματοδότηση να εξασφαλίσει το ότι το σύστημα, η λειτουργία εμπορική βελτιώνεται όταν έχουμε τους διαδρόμους, όταν δεν έχουμε την πολυμορφία, την πανσπερμία που υπήρχε και αυτά έχουν σχέση με τα προγράμματα δράσης. Και τελικά έτσι πιστεύουμε ότι το το οποίο βασικά είναι τα διαβήματα που έχουμε συμφωνήσει με κατασκευαστές, με διαχειριστές υποδομών. Αυτά τα βήματα πρέπει να γίνουν ούτω ώστε το συνέδριο ότι οι κατασκευαστές έχουν συμφωνήσει ότι θα πρέπει να έχουν αυτές τις on-board units συστημάτων προσπαθούμε να υπάρξει διόρθωση όπου υπάρχουν λάθη αφού αυτά τα λάθη. Έτσι η διαδικασία να είναι πιο στεγανή. Τέλος, όσον αφορά την χρηματοδότηση, συνεργαζόμαστε στην με τα για να ευθυγραμμιστούμε όσον αφορά το ΣΕΦ και την χρηματοδότηση και όσον αφορά τη διακοπή κάποιων προγραμμάτων ή έργων έχουμε αυτά τα συστήματα ασφαλείας τα οποία δεν θέλουμε να τα σωρεύσουμε με τα προηγούμενα όπως είχε συμβεί στην Δανία Βέλγιο και Λουξεμβούργο τώρα επίσης προγραμματίζουν να σταματήσουν κάποια παλιά συστήματα και οι κάτω χώρες προς τα εκεί θα κινηθούν άρα έχουμε σημειώσει πρόοδο και αν δείτε τα συμπράσματα του Συμβουλίου έχουν ενθαρρυνθεί όλα τα κρατημέλη να εγκαταλείψουν κάποια παλιά συστήματα οπότε κάποιοι έχουν επενδύσει σε καινούργια συστήματα και μέσω πρόθεσμα προς τα εκεί θα κινηθούν οι περισσότεροι. Νομίζω ότι ολοκλήρωσε και άλλωστε εξήγησε για το χρόνο που μου δώσατε άρα να βάλω ε, εδώ μια τελεία και ευχαριστώ να σας ε, απαντήσω ερωτήσεις για το τι περιλαμβάνει το πρόγραμμά μας αλλά και να συζητήσουμε τα όσα περιέχονται στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Θα επανήλθουμε η κυρία Φίτς και σας ευχαριστούμε. Τώρα να δώσουμε το λόγο. Μην έχετε το λόγο για λίγα λεπτά. Ευχαριστώ για την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Προσωπικά είμαι μεγάλη οπαδός του ERTMS, διότι πια στον 21ο αιώνα θεωρώ ότι πρέπει... Προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχω να πω το εξή. Κοιτάξτε, με... προ... προκαλέσετε κάποια σύγχυση. Πρώτον, το ERTMS κρίνουμε και με πολύ αυστηρή ματιά. Προ λίγων ημερών συναντήθηκα με την κυρία Βένερ και τον κύριο Βίκ από την Επιτροπή και αντίθετα αυγήκε το ελεγκτικό συνέδριο όταν λέει ότι το σχέδιο ανάπτυξης του 2009 έχει στην ουσία αποτύχει. Φυσικά και ανεφάρμοστα. Ακόμη χειρότερα αν γνωρίζει κανείς ότι το 2016 εξοπλίστηκαν με ERTMS μόνο τέσσερις οι άλλοι εκπρόσωποι της Επιτροπής τι είναι αυτό που κάνει τούτο εδώ το καινούριο σχέδιο καλύτερο από το παλαιό. Είναι πιο ρεαλιστική η στόχη μέχρι το 2023. Ε, όπως είπατε εσείς, υπάρχει πλέον η δεσμευτική έγκριση από πλευράς χωρών μελών, ότι δηλαδή θα το ε, υλοποιήσουν. Το πρόβλημα που έχω είναι ότι ο χρόνος εφαρμογής του project δεν συμπίπτει με το χρόνο διάρκειας του πλαισιού χρηματοδότησης. Για το 2007 ε, ε, project βεβαίω και φέρει μέρος της ευθύνης κάθε χώρα μέλος εφόσον δεν απορροφά τα κονδύλια, αλλά 50% των κονδύλων να επιστραφούν είναι πάρα πολλά. Και τώρα, πάλι δεν έχουν απορροφηθεί και για την επόμενη περίοδο επαρκή ε, ε, η περήφανη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που τα κονδύλια επιστρέφουν τουλάχιστον στην διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη. Μπορεί όμω κανεί να μα εγγυηθεί ότι τα χρήματα αυτά, τα κονδύλια αυτά θα επενδυθούν στην ανάπτυξη και εξέλιξη του συστήματος ERTMS στο μέλλον. Υποβάλλει μου φαίνεται λογικό. Ρωτώ τώρα τον κύριο Βίνκ, τι είναι τι έχει βελτιωθεί, γιατί θεωρείτε ότι τα πράγματα βελτιώνονται και ότι ξαφνικά θα συμμετάσχουν όλες οι χώρες και ότι θα είναι επιτυχές. Ρώτησα αυτά τον εκπρόσωπο της ε, Επιτροπής, κ. Βίνκ. Μου απάντησε, «Λοιπόν, είμαι αυστριακή όπως θα έχετε καταλάβει και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρώ ότι πρέπει να διδαχθεί από την μη η ιδεώδη ή τιμή μη ιδανική ε, επίλυση των θεμάτων του παρελθόντο, το, το ERTMS. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και γιατί με τις συμφορά προσώπια τη παρουσιάσεω τώρα. Προ 14 ετών ήμουν εισηγητή για το ERTMS. Και τα είχαμε ήδη συζητήσει όλα αυτά τα πράγματα τότε. Θα σας πω ότι 14 χρόνια δεν εγγνωμούμε πολλά εκατομμύρια και στην ε, σηματοδότηση αλλά και στην συντήρηση των σηματοδοτών. Και γίνεται πάντα επενδύσει στην υποδομή μόνο εφόσον θεσπίσουν το ERTMS. Και τίποτα δεν έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το δεύτερο είναι ότι οι εγωισμοί των χωρών μελών ήταν τόσο ισχυροί <clears throat> ώστε το ERTMS να το αλλάζουν διαρκώς. Ώστε να έχουμε και δεν είναι το ζήτημα ότι δεν έχουν αρκετά για τη συγχρηματοδότηση, δεν απορροφούν ούτε τα κονδύλια. Και όταν μιλήσαμε για 50% για το retrofitting, αυτό ισχύει διότι η υψηλή δηλαδή συγχρηματοδότηση από την Ευρώπη, διότι είναι διαμεθοριακό ε, σχέδιο. Εγώ Απαγορεύτηκε μεν στις χώρες μέλη να ανανεώνουν τα διαφορετικά τους παλαιά συστήματα, αλλά ούτε αυτό βοήθησε τίποτε, διότι τελικώ τα συμφέροντα της βιομηχανίας και εθνική εγωισμή ήταν μεγαλύτερη από την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Πρέπει να μην δώσει χρήματα πλέον στις χώρες μέλη για τις υποδομές, εάν δεν δεσμευτούν για την πλήρη χρήση του ERTMS και γιατί θα κάνουν για συγκεκριμένες συνδέσεις. Η Deutsche είχε διαπραγματευτεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα ήταν από τη συνολική απόσταση των 150-200 χιλιόμετρων τα 30 χιλιόμετρα δεν είχαν διερθεί εμεί και για το λόγο αυτό είπε η Deutsche Bahn, α, δεν θα το κάνουμε. Δεν με ενδιαφέρουν πλέον οι διατυπώσεις, οι φραστικές διατυπώσεις, με ενδιαφέρουν τα γεγονότα. Καλά, λαμβάνει, λαμβάνει δισεκατομμύρια για ορισμένα project. Για παράδειγμα, Στουτγάρδη, 10 δισεκατομμύρια για να γλιτώσουν λίγα λεπτά διαδρομής. Τελευταίο, εκτός από τη Δανία υπάρχει και άλλη μια χώρα που τα έχει καταφέρει να το αναπτύξει σε όλη την επιφάνεια. Το καταφέρνει η Ελβετία διότι είναι τόσο ευρωπαϊκή που δεν χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε. Το ελεγκτικό συνέδριο πρωτίστως για την εξαιρετική αυτή έκθεση. Ας μην γελιόμαστε ωστόσο διαβάζει κανείς ανάμεσα στις γραμμές στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου κριτική κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και εδώ θα συμφωνήσω και με, λέμε καμιά φορά, πίνετε ένα ποτήρι μπύρα, κάνετε λίγο πιπί και τα πράγματα είναι πάλι ίδια. Δηλαδή στην ουσία αυτό μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Αυτό οφείλω να ομολογήσω στην ε, στην αγορά το iPhone με τον ίδιο τρόπο που πάει να πουλήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ERTMS, θα καθόμασταν ακόμα με κάποια απαρχαιωμένα τηλέφωνα στα χέρια. Ούτε και το ERTMS είναι το iPhone. Αλλά καταφέραμε ορισμένα πράγματα να τα προχωρήσουμε πολύ γρηγορότερα από τη δέσμευση από πλευρά χωρών μελών. Εγώ δεν την βλέπω. Προ 1,5 έτους έγινε στη Γερμανία ένα βαρύ ατύχημα. Καταστράφηκε μια σύραγγα και χρειάστηκε να κινηθούν τα τρένα μέσω Γαλλίας. Αδύνατον. Διότι ότι κάθε μια χώρα μέλους κάνει τα δικά της. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται πολιτική συζήτηση και θα το προτείνω στον γύρο των συντονιστών όπου θα προσκληθεί η Επίτροπος. Αν καθίσουμε τώρα να δούμε ποιες διαφορές υπάρχουν, βλέπουμε ότι δεν λειτουργεί τίποτα. Ενώ δαπανώνται ότι το ERTMS είναι πραγματικά όριμο τεχνικά. Γιατί το ρωτώ αυτό. <clears throat> Κάπως με ενοχλεί το εξής. Προ εβδομάδων ανοίξαμε μία διαδρομή 600 χιλιόμετρων για ε, υψηλή ταχύτητα και από ό,τι λένε οι εφημερίδε, οι δυσκολίε που σημειώνονται εκεί, οι διαρκεί διακοπέ, πάρα πολλέ δεκάδε διακοπών, για αυτέ ευθύνεται το ΙΕΤ. Ναι, ότι τα πράγματα είναι δύσκολα για να αξιολογηθεί το κόστο. Και θα πρέπει να διαπιστώσουμε το ότι τα, κάποια συστήματα ασφάλειας, κάποια κατημέλη πρέπει να υπάρξει αντικατάσταση γιατί έχουν παλιώσει. Και να δούμε σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να γίνουν κάποιες δαπάνες οι οποίες όμως θα γίνουν για να μπει το ERTMS αλλά έχουμε λιγότερο από χίλια χιλιόμετρα από τα 30.000 που ισχύει το ERTMS όμως έχουμε πριν από το ERDMS έχουμε σε ένα κράτος μέλος τρία διαφορετικά συστήματα ε, σηματοδότησης. Βλέπουμε ότι υπάρχει δυσκολία από πλευράς χρηματοοικονομικής. Επίσης κύριε Μπάλκο, θα εξηγήσουμε πώς θα αναδείξουμε το όφελος του συστήματος από πλευρά οικονομικής πάντα. Είπαμε για καλύτερη ταχύτητα, πυκνότητα κυκλοφορίας θα έχουμε απόδοση των επενδύσεων. Καλά με τις ενισχύσεις και τις επιδοτήσεις. Μπορούμε να έχουμε όμως οικονομικά κίνητρα. Γιατί αν δεν υπάρχουν καλά με τις ενισχύσεις και τις επιδοτήσεις. Μπορούμε να έχουμε όμως οικονομικά κίνητρα. Γιατί αν δεν υπάρχουν αποδόσεις από τις επενδύσεις, για ε, τα πράγματα δυσκολεύουν. Άρα θα πρέπει να δούμε τι δαπάνη υπάρχει και αυτές οι δαπάνες πώς αποσβαίνονται. Και όσον αφορά τον κύριο Φίτς, την Επιτροπή, για την υποδομή. Είναι θέμα του κράτους παντού. Και το πρόβλημα αυτών των διαφορετικών συστημάτων σηματοδότησης δεν αναφέρεται αρκετά ούτε από τους πολιτικούς ούτε από τα μέσα ενημέρωσης. Και ακριβώς από το ότι φτιάξαμε μια υπηρεσία να ρυθμίσει τα των ιδιομορφιών των διαφορών δρόμο επίδειξης από το Ρότερνταμ. Αυτό έχει προχωρήσει. Οπότε να δώσουμε για να, και μετά να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις... Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, όπως είπατε στην αρχή, αλλά και στην τωρινή σας παρέμβαση. Η έκθεση αυτή παρουσιάζει την, τις τα τεχνικά, τα οικονομικά ζητήματα και τα ζητήματα υποδομών Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την κυρία Σμίτ για το σε επίπεδο κοκομπού, ε, ελέγχου των προπολογισμών, όταν ε, παρουσίασα την έκθεση αυτή. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, κυρίως για τις ε, οικονομικές πτυχές ε, του όλου θέματος και βάσει αυτή τη συζήτηση μπορούμε να δούμε ότι έχουμε δίκιο σε αυτά που λέμε στην έκθεσή μας. Δεν ήμασταν μόνο επικριτικοί, ήμασταν και επικοδομητικοί. Παρουσιάσαμε την ενδεχόμενη κατεύθυνση της ανάπτυξης αυτού του σημαντικού εγχειρήματος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει επίσης και το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, το έγγραφο εργασίας που ε, αναφέρεται στο πώς, ε, ποια θα είναι η πορεία μας στο μέλλον. Αναφέρεται σε κάποια προβλήματα που εντοπίζονται και στο δικό μας και στη δική μας έκθεση. Κοιτάξτε, εμεί δεν είμαστε τεχνικοί, ελεγκτές είμαστε και είμαι ας πούμε συγκρατημένα αισιόδοξο. Αν μέσω της συζήτησης αυτής μπορούμε να δούμε ότι είναι ενδιαφέρον για την Επιτροπή σας και επειδή είπε και ο κύριος Κράμερ, τόνισε μάλλον ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε ε, και πριν ε, από 14 ε, χρόνια το θέμα αυτό και είναι πολύ αργή η πρόοδος. Αν λοιπόν συμφωνείτε, εμείς μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα μετά από λίγο καιρό και να προετοιμάσουμε μία παρακολούθηση, ένα follow-up, μία συνέχιση μάλλον της, της παρακολούθησης κατάστασης από εμά και να δούμε πώς θα, τι πρόοδος θα σημειωθεί. Και θα ήθελα να ζητήσω και από τον κύριο Ούλμπανιτς που συμμετείχε στην ε, έκθεση αυτή να προσθέσει και εκείνος κάτι αν θέλει. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συμπληρώσω αυτό που είπε μόλις ο κύριος Μπάλκο για να απαντήσω λίγο καλύτερα στην ερώτησή σας. και σε σχέση με τα ερωτήματά σας. Εμείς προσπαθήσαμε στην έκθεσή μας να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ της μεμονωμένη ας πούμε, ε, οικονομικής αποδετικότητας για κάθε φορέα και της Ευρωπαϊκής Ένωση, όπου εκεί δεν υπάρχει καμία ε, αμφιβολία. Αν καταφέρουμε να είμαστε πιο πιστικοί για τους φορεί εκμετάλλευσης ω, προ... Ε, χρηματοδοτηθεί κιόλα. Θα είναι πιο εύκολο δηλαδή να φέρει κανείς το βάρος της, ε, του κόστους ε, που ε, του αναλογεί. Δεν είναι πολύ εύκολο αν είμαστε λοιπόν πιο πιστικοί ως προς αυτό το κομμάτι και μπορέσουμε να πείσουμε τους φορείς εκμετάλλευση για θελοντικά ε, στην όλη διαδικασία τι τέτοιο να ενθαρρύνει ε, δηλαδή τους φορείς εκμετάλλευση, ποια είναι τα πλεονεκτήματα που μπορούν ε, να δουν γιατί θα, θα θέλαμε και εμεί και τα κράτη-μέλη και οι Ευρωπαϊκοί πιστούν ότι αξίζει τον κόπο διότι βεβαίω η επένδυση είναι βραχυπρόθεσμη σε βάθος χρόνου κερδίζουν και πολλοί. Ε, ήταν μεμονωμένοι, ο καθένας δηλαδή δούλευε μόνος του και δεν υπήρχε η απαραίτητη συνεργασία με το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο τώρα. Έχουμε ε, συγκεκριμένες αρχές, επίπεδο κράτους μέλους, πρέπει να υπάρχει μια, ένα συντονισμός τη διαχείριση του στήματος και είναι πάρα πολύ σημαντικό και το εξή ότι έχει ένα ρόλο στην έγκριση κάθε νέας, ε, κάνει ένα πρόγραμμα σε εθνικό επίπεδο, να αναπτύξει το πρόγραμμα σε, εθνική, σε εθνικό επίπεδο πρέπει να περάσει περάσει μέσα από τον ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό ε, Σιδηροδρόμων, τον ERU. Υπάρχει μια ε, μεθοδολογία η οποία ελπίζουμε ότι θα είναι αποτελεσματική ως προς το κόστος. Καταλαβαίνουμε την απογοήτευση των καταναλωτών. Κάνουν μια προσπάθεια επανεξοπλισμού γιατί καταλαβαίνουν ότι το ευρύτερο σύστημα είναι πιο επωφελές το σύγχρονο ERTMS ε, του και για τους φορείς εκμετάλλευσης. Αυτό είναι σημαντικό. Ε, και η ομάδα ανάπτυξης μας ε, δουλεύει προς αυτό για να δείξει δηλαδή ότι η οικονομική αποτελεσματικότητα του ERTMS έχει σχέση και με αυτό. Δηλαδή είναι κάτι που είναι σημαντικό και για τους φορείς εκμετάλλευσης. Να πείσει δηλαδή τα κράτη-μέλη ότι είναι μια επένδυση που έχει νόημα που έχουν γίνει από τους φορείς εκμετάλλευσης των κρατών μελών δείχνουν ότι ο ε, ότι ο γερμανικός διάδρομος θα είναι ε, σύντομα πλήρως ε, λειτουργικός και γι' αυτό ακριβώς τα διασυνοριακά κομμάτια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε επίσης και κράτη-μέλη τα οποία ε, τα οποία μας υποβάλλουν κάποια συστήματα εθνικής ε, υλοποίησης, εφαρμογής του συστήματος ε, και ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε σε μια λειτουργία και των εθνικών σιδηροδρόμων που θα βασίζεται αμυγός στο ERTMS. Σε σχέση με αυτά που είπε ο ERT, το, κύριος Κράμερ, είναι σημαντικό όλο το τροχαίο υλικό να έχει, τουλάχιστον επί του σιδηροδρόμου, να υπάρξει αυτή η προδιαγραφή 3 η οποία θα ισχύει σε όλες τις μονάδες επί του σιδηροδρόμου και που πρέπει να είναι συμβατή με όλο το RTMS όπως έχει αναπτυχθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο κύριος Κόχας έθεσε το θέμα της νέας ταχείας στη Γερμανία. Πράγματι, αυτό ήταν μια καταστροφή για την Deutsche Bahn. Ε, Βεβαίω την εξετάσαμε για προφανείς λόγους, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα λόγω του ERTMS. Απλώς ήταν, ήταν λάθος οι παράμετροι του συστήματος, ε, ε, ήταν διαφορετικό το μέγεθος των τροχών σε, κάποιες, ε, σε κάποιους σειρμούς και δεν είχαν εκπαιδεύσει σωστά κάποιους από του οδηγού σε σχέση, οδηγούς σε σχέση με το σύστημα τροχοπέδησης των σιδηροδρόμων. Για την ώρα πάντω όλα πάνε καλά και χαίρομαι όλου ιδιαίτερω. Κύριε Βαντερκάμπ, θέσατε το ευρύτερο ζήτημα ε, που υπήρχε στον, στο διάδρομο Ρότερνταμ ε, Reichstag στη Γερμανία πέρσι είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα ε, γιατί έπρεπε να περάσουν ε, οι εμπορευματικές μεταφορές από τη Γαλλία. Μιλήσατε ορισμένοι εξημών από τα, για τα ζητήματα διαλειτουργικότητας. Υπήρχαν θέματα που τα γνωρίζαμε, αλλά το συγκεκριμένο θέμα, η συγκεκριμένη υπόθεση μας έδειξε και σε εμά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πρόβλημα. Ε, μας το έδειξε δηλαδή καθαρά το πρόβλημα της γλώσσας, το πρόβλημα της εκπαίδευσης των οδηγών. Ε, πραγματικά ζητήματα τεχνικής διαλειτουργικότητας και αναγκαστήκαμε να, βρούμε, να προσπαθήσουμε να βρούμε τα, τα, λύσεις, ε, τουλάχιστον τις λύσεις που ε, μπορούμε σε πρώτη φάση να εντοπίσουμε για να λύσουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Για το, το συνδέοντα την Ευρώπη. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε το εξή. Παρά το γεγονό ότι υπήρχαν ε, πολύ μεγάλα επίπεδα ε, ε, μάλλον πρόβλεψης εκταμιεύσεων ε, για το διάστημα 2014 με 2016. Δεν έγινε όμως κάτι τέτοιο. Η ταχύτητα με την οποία θα χρηματοδοτούνταν τα projects δεν ήταν κάτι που μπορέσαμε να τηρήσουμε. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε τώρα έναν καλύτερο κανόνα. Η ότι περιμένουμε περισσότερο να προχωρήσουν τα projects ε, μέχρι να ε, δεσμευτούμε ως προς τα ποσά που θα διατεθούν. Έτσι προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε. Όσον αφορά λοιπόν τη σταθεροποίηση του ERTMS, ε, την μεγαλύτερη διαθεσιμότητα, την εμπορική του συστήματος, το θέμα των προδιαγραφών, των νέων προδιαγραφών είναι κάτι το οποίο είναι σχετικά πρόσφατο και ελπίζουμε ότι σε δύο-τρία χρόνια θα ξανασυζητήσετε το πρόβλημα αυτό και ελπίζουμε μέχρι τότε να δούμε την πρόοδο που ε, θα διαπιστώσετε κι εσείς ε, και την πρόοδο που χρειαζόμαστε για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά το Ιαρίστος ε, να μας Επισκεφτείτε και πάλι να μας παρουσιάσετε τη δική σας εκτίμηση για την κατάσταση. Πάντως είναι να ζητώ λοιπόν πάρα πολύ κύριε Φίτς, Μπάλκο και την ομάδα σας ε, που ήρθατε να μας ε, παρουσιάσετε τις εκθέσεις σας. Συνδυασμένες μεταφορές. να δώσουμε πρώτο το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατόπιν να ακούσουμε την κυρία Γιούτο που είναι η συγγετρία και κατόπιν να ακούσουμε τους σκιώδες συμπάτου. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε που μας δίνετε την ευκαιρία να σας ε, παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας για αυτή την ε, οδηγία που αφορά τις συνδυασμένες μεταφορές. Για να δούμε τώρα τις ε, ε, διαφάνειές μας πρώτα-πρώτα για να δούμε λίγο το πλαίσιο αυτής της πρότασής μας. Εντάσσεται σε κάποιες πρωτοβουλίες οι οποίες ε, κοπούν στο να προχωρήσει η υπόθεση των συνδυασμένων μεταφορών. Βλέπετε τώρα πώς έχει η σημερινή κατάσταση, πώς κυριαρχούν στις μεταφορές οι οδικέ μεταφορέ ε, φορτίου που είναι περίπου το 50%. Εάν κανεί μπορούσε να αυξήσει τι συνδυασμένε μεταφορέ θα υπήρχαν πολλέ θετικέ συνέπειε όσον αφορά την μείωση των βλαπτικών εκπομπών γιατί τα τρία τέταρτα αυτών προέρχονται τι οδικέ μεταφορέ σήμερα. Επίση, θα είχαμε θετικέ συνέπειε και όσον αφορά την ασφάλεια γιατί τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν στου δρόμου. Επίσης πλεονεκτήματα και για την ε, ατμόσφαιρα και επίσης θα είχαμε πιο ισόρροπη χρήση των δικτύων μεταφοράς. Γιατί σήμερα ε, έχουμε ε, πάρα πολύ χρήση των δρόμων και το οικονομικό κόστος είναι βαρύ. Για να δούμε τι θα πει συνδυασμένη μεταφορά. Πρόκειται για κάποιο είδος πολυτροπικών μεταφορών και εννοούμε τις μεταφορές που χρησιμοποιούν ένα κοντέινερ που έχει κάποιο φορτίο και αυτό το κοντέινερ πηγαίνει από ένα τρόπο μεταφοράς σε κάποιον άλλο. Επίσης με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε το κομμάτι της διαδρόμης που χρησιμοποιούν τρόπους μεταφοράς εκτός δρόμου. Ο δρόμος επομένως είναι η αρχή και το τέλος της διαδρομής. Συνδεσμένη μεταφορά είναι υπόθεση που πάει καλά τελευταία. Καλές είναι οι επιδόσεις, αλλά θα μπορούσαμε να πάμε ακόμα καλύτερα. Άρα για να δούμε ποιο είναι ο λόγος που δεν βλέπουμε να χρησιμοποιούνται περισσότερο συνδυασμένες μεταφορές. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλε υποδομές, να υπάρχει ε, τρόπος της μεταφόρτωσης από το ένα μέσο μεταφοράς στο άλλο σε μερικά μέρη στην Ευρώπη υπάρχουν τέτοιες ε, διευκολύνσεις, αλλά αλλού δεν υπάρχουν. Χωρίς να υπάρχει ομένω τέτοιου είδους διευκόλυνση, τέτοιου είδους τρόπος δεν υπάρχει συνεσμένη μεταφορά. Για να δούμε, μείνουμε σε αυτή τη διαφάνεια, γιατί είναι και το θέμα των δαπανών. Βλέπετε εδώ κάποιες ε, εκτιμήσεις για την μέση μεταφορά φορτίου για κάποιες αποστάσεις 500-600 ε, χιλιόμετρων. Εάν 100 είναι το κόστος να χρησιμοποιήσει κανείς μόνο τον δρόμο, η συνέσμενη μεταφορά χωρίς ε, κάτι άλλο ε, επιπλέον παρέμβαση όπως είναι 25% παραπάνω. Οπότε, εάν έχουμε κάποια κλασική καθαρή μορφή μεταφορά, να έχουμε κάποιε εξοικονομίες, να έχουμε επομένω μόνο γιατί φορτηγίδε, δρόμο μόνο σε δρόμο λοιπά, Αλλά όλες αυτές οι οικονομίες εκμυδενίζονται από την ε, δαπάνη της μεταφόρτωσης των κοντέινερ. Αλλά υπάρχει και επιπλέον κόστος. Βλέπετε εκεί στο, στο κίτρινο της επιπλέον δαπάνης Οπότε κανείς θα πρέπει κάτι να ρυθμίσει με περισσότερους ε, εμπόρους, περισσότερους παρόχους και οπότε υπάρχουν και άλλα θέματα πια αξιοπτήρες οπότε έχουμε και άλλες δαπάνες. Τις δαπάνες που επιβάλλει ε, ο κανονισμός, εάν κανείς δεν κάνει αυτό που πρέπει. Τι εννοώ με κόστος από τον κανονισμό. φέρει Φερρυπίν υπάρχει ε, ένας κανονισμός αφορά το βάρος, τις διαστάσεις, τι μπορεί να μεταφερθεί. Αλλά στις συνεργασμένες μεταφορές έχουμε ένα βαρύ κοντέινερ και έτσι μειώνεται το βάρος μπορεί κανένας να βάλει επιπλέον να μεταφέρει. Άρα και αυτό σημαίνει ε, δαπάνη, κόστος. Ε, το βάρος μπορεί κανένας να βάλει επιπλέον να μεταφέρει. Άρα και αυτό σημαίνει ε, δαπάνη, κόστος. Ε, ε, Καμποτάς τώρα. Αν κανένας χρησιμοποιήσει μόνο τους δρόμους στη διεθνή μεταφορά, τότε δεν ισχύουν αυτές οι διατάξεις. Αν κάποιος όμως δεν κάνει το ίδιο με τη συνδεσμένη μεταφορά, έχει καμποτά τώρα. Αν κανένα χρησιμοποιήσει μόνο του δρόμου, στη διεθνή μεταφορά, τότε δεν ισχύουν αυτέ οι διατάξει. Αν κάποιο όμω δεν κάνει το ίδιο με τη συνδεσμένη μεταφορά, έχει. Η οδηγία ανάγεται στο 92, είναι παλιά, θέλει επικαιροποίηση. Αλλά πιο συγκεκριμένα πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε τα θετικά. Άρα θα πρέπει να στραφούν όλοι στο δρόμο. Ε, τώρα για να δούμε θα πρέπει να είναι πιο ξεκάθαρος ο ορισμός. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρος ε, όπως έχει σήμερα η νομοθεσία. Ορισμός του διασμένης μεταφοράς. Έχουμε μεγάλη αβεβαιότητα επομένως από πλευράς ε, των εμπλεκομένων τη συνδυασμένη μεταφορά πολλές φορές χρησιμοποιείται σαν πρόφαση για να παρακάμψει κανείς τον νόμο παρακάμψει στις διατάξεις του καμποτάζ. Αυτό βέβαια είναι ανεπιθύμητο. Θέλουμε και έτσι να εξασφαλίσουμε ότι οι μεταφορές είναι ε, ολογίες για κάποια έγγραφα έτσι θα μειωθεί το διοικητικό άχθος για τους μεταφορείς. Επίσης θέλουμε να επικαιροποιήσουμε τα κίνητρα που έχουν σχέση με τις μεταφορές. Για να δούμε τώρα. Να δούμε τις λεπτομέρειες περισσότερο όσον αφορά τον ορισμό. Ο πιο κοντινός, ο πιο δόκιμος, γιατί αυτό οδηγεί σε παρερμηνίες, οδηγεί σε ένδικες διαφορές, προστριβές και άρα να πάμε σε κάτι απλούστερο ως οδηγό και οι αρχές έτσι να μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα. Βλέπετε εδώ αυτές τις λεπτομέρειες. Άρα θέλουμε να συσχετήσουμε κάποιο είδους ε, στοιχεία, πληροφορίες που θα πρέπει να δίνονται περισσότερα από όσες σήμερα να μπορούμε και εμείς να επαληθεύσουμε ότι η μεταφορά η συγκεκριμένη αποτελεί συνδυασμένη μεταφορά παροχή αυτών των στοιχείων και πληροφοριών. Και το καλό είναι πιο εύκολο οι αρχές να διαπιστώνουν αν υπάρχει συμμόρφωση με τον νόμο. Άρα όλα θα δεινά η ILU για τα containers σε όλη τη διάρκεια της μεταφοράς. Τέλος. Όσον αφορά τα κίνητρα. Όπως είπαμε προηγουμένως, η μεταφορά έχει έτσι κι αλλιώς οδηγία να υπάρχουν δηλαδή παντού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση κατάλληλε και απαραίτητε υποδομέ για τη μεταφόρτωση, για τι διευκολύνσει που υπάρχουν ε, σε κάποια μέρη, αλλά όχι παντού. Αλλού λείπουν. Οπότε με αυτή την πρόταση πρώτα-πρώτα θέλω, αλλά θα αφαιθεί το περιθώριο στα κρατημέλη αποφασίσουν τι θα κάνουν, γιατί οι συνθήκες διαφέρουν από τη μια χώρα στην άλλη. Οπότε τα κρατημέλη θα πρέπει να παρέμβουν ούτως ώστε να βοηθήσουν με τις διευκολύνσεις της μεταφόρταφορας. Της μάλλον. Τώρα πάμε στην τελευταία διαφάνεια. Βλέπετε το αποτέλεσμα κάποιων simulations που κάναμε προσωμιώσεων δηλαδή. Οπότε, εάν Οπότε είδαμε ότι έτσι θα έχουμε 17% αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Δηλαδή το πόσο θα ωφεληθεί ο κλάδος. Τώρα δημοσιονομικά ωφέλη για τα κρατημέλη. Λογικά. Αύξηση της ε, αλλαγής ε, της χρησιμοποίησης τέλο πάντων περισσότερων τρόπων μεταφοράς κυρίως για τις μεγάλες αποστάσεις και όπως είπαμε και στην πρώτη διαφάνεια πρόκειται οι επιπλέον δαπάνες να περικοπούν και σας... που είναι η συγγήτρια για... αισθάνθηκα υπερήφανη γιατί αυτές οι μεταφορές αυτός ο τρόπος μεταφοράς είναι αυτό το οποίο πρεσβεύει η πολιτική μας ομάδα. Θεωρούμε ότι έτσι θα πρέπει να γίνονται οι ευρωπαϊκές μεταφορές, η συμφόρηση στους δρόμους. Άρα περήφανοι που το ανέλαβα ήταν πολύ καλή συνεργασία με τους ε, συναδέλφους και η πρόταση του Κοινοβουλίου θα πρέπει να προσεγγίζει όσο γίνεται περισσότερο σε κάποια λύση που να... δεν την αλύσαμε στις λεπτομέρειες σήμερα. Αλλά εμείς είπαμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό, πολύ είναι θετική, γιατί μιλούμε για επικαιροποίηση της νομοθεσίας του 92 και δεν είναι μόνο θέμα μεταφοράς. Είναι ε, θέμα το τότε. Ήταν θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να πάμε καλά για τους στόχους που έχουμε. Δηλαδή, πρώτα-πρώτα προστασία της υγείας, προστασία του περιβάλλοντος. Όλοι μας συμφωνούμε όσον αφορά το ότι θα πρέπει αυτοί οι στόχοι να επιτευχθούν. Άρα να δούμε τις επιπτώσεις των μεταφορών επί υγείας και επί του περιβάλλοντος. Δηλαδή, να εγκαταλείψουμε του μολυσματικούς, τους ρηπαντικούς τρόπους μεταφοράς όπως η οδική μεταφορά. Πάμε σε πιο καθαρές μεταφορές. Άλλο πολύ βασικό και γι' αυτό θα ωφελήσουν οι συνδυασμένες μεταφορές είναι εξυγχρονισμός από συμφόρηση όσον αφορά τα logistics την επιμελητεία. Γιατί τώρα τελευταία έχουμε δει μεγάλες αλλαγές. Θα πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε, να εξυγχρονίσουμε όλο τον τομέα των μεταφορών από συμφόρηση Επομένω των οδικών μεταφορών χρησιμοποιούνται άρα να δούμε πώ θα μπορέσουμε να γεφυρώσουμε αυτές τις διαφορές που υπάρχουν λοιπόν προβλήματα στην Ευρώπη στα δίκτυα αλλά και στα hubs, στους κόμβους Λοιπόν, προβλήματα στην Ευρώπη στα δίκτυα αλλά και στα hub, στους κόμβους. Άρα η πρόταση του Κοινοβουλίου και ελπίζω να συμφωνείτε μαζί μου κατατείνει στο ότι θα πρέπει να γεφυρώσουμε τις διαφορές από τόπο σε τόπο στην Ευρώπη. Αλλιώς πώς να προωθήσουμε τους τρόπους μεταφοράς που θέλουμε. Αλλιώς θα είναι το κόστος υυξημένο και ο κόσμος θα ξαναελκύεται από τις οδικές μεταφορές. Θα πρέπει οι οι αλλαγές να συνοδεύονται από κάποια πλεονεκτήματα διαφόρων ειδών και άρα οι εταιρείε μεταφορών και τα κράτη να ελκύονται από την πρότασή μας και να πηγαίνουν προς τα εκεί που θέλουμε. Να βρούμε επομένω το πώς οι βασικές ε, δαπάνες, το κόστος που συνεπάγονται θα ε, δικαιολογεί την, την, την αλλαγή, τη στροφή. Πέραν, είπαμε, το, το, το, το για την υγεία κλπ. Και όλα αυτά θα πρέπει να αφορούν και τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Τώρα για τα ψηφιακά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφάνεια και τα ψηφιακά. Θα είναι πιο γρήγορος ο έλεγχος, ο αδύνατος κρίκος των μεταφορών και κυρίως στο, στο δρόμο των οδικών είναι ο έλεγχος. Δύσκολο να γίνουν όσοι έλεγχοι χρειάζεται, αλλά και αυτοί που γίνονται συνεπάγονται αυξημένη γραφειοκρατία. Επομένως, δεν θα πρέπει τα μειονεκτήματα, οι δυσκολίες του ελέγχου να αποτελούν αντικίνητρο και άρα ο κόσμος να φεύγει από έναν τρόπο μεταφοράς που θέλουμε. Χρειάζεται διευκόλυνση, χρειάζεται κατάργηση γραφειοκρατίας και να προσέξουμε την αύξηση του κόστου, την αύξηση των δυσκολιών για τους τρόπους μεταφράσεων που θέλουμε να προωθήσουμε. Για να δούμε τώρα τις λεπτομέρειες πρότασης της Επιτροπής. Να ξεκινήσουμε με το θέμα του ορισμού. Άρθρο 1 δηλαδή. εξηγήθηκε γιατί θα πρέπει να είναι ο ορισμός πιο σαφής. Έχουμε αυτά τα 150 χιλιόμετρα, έχουμε αυτό το 20% εκτός δρόμου κλπ. Αυτό είναι, είναι κριτήρια που φέρνουν περισσότερη σαφήνεια. Να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε ε, προβλήματα σε σχέση με τον ορισμό. Και όπως έχουμε πει και σε άλλη συζήτησή μας, να προσέξουμε πως αυτή μας η πρόταση θα οδηγήσει σε αποκλήσεις προβληματικές, σε αντιφάσεις με άλλες οδηγίες. Αναφέρθηκε ας πούμε η νομοθεσία για βάρος και διαστάσεις σε αυτό θα πρέπει να προσέξουμε όσον αφορά τον ορισμό. Πάντως, θεωρούμε θετικό το ότι στον ορισμό ε, λαμβάνονται υπόψη τα των στάνταρ, των προτύπων. Είπαμε για τους ε, ελέγχους, λέω για το άρθρο 3, είναι πάρα πολύ ειδικές μεταφορές. Και ίσως θα πρέπει να δούμε πώς τα έγγραφα ελέγχουν να χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία έτσι θα πρέπει να μειώσουμε την γραφειοκρατία έτσι το σύστημα έλεγχο την υποβολή εκθέσεων αναφορών κατά τη γνώμη μας η πρόταση της Επιτροπής καλά τα λέει ότι τα κρατήμε δηλαδή πρέπει να σαφείς στόχοι ας πούμε μείωση εκπομπών ε, Κυρία Γιούτορ, λέει ο πρόεδρος, θα πρέπει να ολοκληρώσετε, γιατί έχετε υπερβεί τον χρόνο που προβλέπαμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, σύντομα θα τελειώσω. Δύο-δύο σημεία τώρα. Πάρα πολύ σύντομα όσον αφορά το καμποτάζ και την απόσπαση εργασομένων, διότι, διότι λέγω γνωρίζουμε ότι για τις συνδεσμένες μεταφορές το κομμάτι που είναι οδική μεταφορά την χάνει εξαίρεσης, παρέκκλησης για το καμποτάζ. Δεν ισχύει και το καμποτάζ, οπότε να προσέξουμε. Να μην το εκμεταλλεύονται αυτό οι εταιρείε για να παρακάψουν τον νόμο μια που δεν ισχύει κανείς το καμποτάζ. Και για την απόσπαση των εργαζομένων θα πρέπει για συνδεσμένες μεταφορές να υπάρξει ρύθμιση ε, από το κοινωτικό δίκαιο και συγγνώμη. Τρία λεπτά. Ε, να αρκεστείτε σε τρία λεπτά για να μπορέσουμε να κάνουμε μια καλή συζήτηση και μετά να εξετάσουμε και το επόμενο θέμα για να έχουμε χρόνο. Κυρία Σμίτ από το ΕΛΚ, τρία λεπτά έχετε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στατιστικές. Βλέπει κανείς εκεί ότι οι μεταφορές δεν μπορούν να σχεδιαστούν κεντρικά. Έχουμε ρίξει δισεκατομμύρια στο σιδηρόδρομο, θα έπρεπε κανονικά να είχαμε δίκανα. Συμβούλιο Κομισιόν και Ευρωκοινοβούλιο, διότι και οι τρεις θεσμοί δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά των μεταφορέων και των μεταφερομένων ε, με νομοθετήματα. Χρειάζεται καινοτομία. Όταν μιλούμε για και όσο εμείς επιμένουμε στο σιρόδρομο, τόσο περισσότερο πηγαίνουν στα αυτοκίνητα. Και η μεταφορά μέχρι το 2030 το 30% να μετακινηθεί δηλαδή από νερότερος δηλαδή και πιο αργός δεν πρόκειται να επιτύχει αυτό. Ακόμα μάλιστα και αυτοκίνητα σειραγές θα κυκλοφορούν αυτόνομα φορτηγά αυτοκίνητα στους αυτοκινητοδρόμους. Άρα τελικώς όλα αυτά συνηγορούν υπέρ του δρόμου και διερωτώ και από ποια απόσταση και πέρα ε, αξίζει τον κόπο οι Αμερικανοί τα φορτώνουν κατευθείαν στα φορτηγά. Δεν κατευθείαν, συγγνώμη, στους σιδηροδρόμους τα εμπορεύματα. Και ενώ εδώ στην Ευρώπη είναι πρώτα το φορτηγό αυτοκίνητο, μετά ο σιδηρόδρομο, μετά πάλι το φορτηγό. Στρατευτισμό των σιδηροδρόμων στι χώρε μέλη δεν έχουμε πολλέ πιθανότητε να δούμε διατροπικέ μεταφορέ. Θέλετε φθηνότερε μεταφορέ. Και να πω ακόμα πολύ σύντομα, έξω υπάρχει μια θαυμάσια έκθεση του Wim van der Kamp για τι συνδιαμένε μεταφορέ. Μπορεί κανεί εκεί να πάει, να ενδιαφερθεί, να... Έχω κάποιε σκέψει μου θετικές και κάποιες ε, με επιφυλάξεις. Εκεί η διάταξη που λέγει το όχος της ρύθμισης είναι να σταματήσει υπάρχει αβεβαιότητα. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τα κίνητρα, πρέπει να δοθούν το πώ θα υπάρξει από ε, όσον αφορά τι οδικέ μεταφορές. Αυτά θα πρέπει να συνεχιστούν με το βασικό στόχο, δηλαδή θα πρέπει να έρθουν οι αβεβαιότητε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Να σταματήσει επίσης η διάκριση μεταξύ κοντέινερ του ωκεανού και των λοιπών. Από τους φραγμούς που υπάρχουν και έτσι να μπορέσουμε να ευνοήσουμε τις συνδεσμένες μεταφορές. το παραπάνω πάμε στα 250 χιλιόμετρα. Και αυτό θα βοηθήσει στην ερμηνεία της διάταξης. Επίσης προσοχή για το πρόβλημα με το καμποτάζ γιατί δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτή η γκρίζα ζώνη, η ζώνη αυτή η πλεονεκτική και έτσι μέσω της μεταφόρτωσης μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει μια τρίτη χώρα πιο φτηνή και... Ευχαριστούμε κύριε Ντεμόντε. Ο κύριος Ροτόφσκι από το ECR. Τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρους της ομάδα μας, της πολιτικής μας ομάδας, θα ήθελα να σας πω ότι εμείς υποστηρίζουμε την ιδέα της ναθανθεώρησης οδηγίας ε, του 1992. Αυτόν είναι πολύ γνωστά. Δύο παρατηρήσεις έχουμε σε σχέση με πολύ συγκεκριμένες λύσεις. Πρώτη παρατήρηση, επέκταση των κανόνων. Σε... Εμείς βλέπουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα στο μέλλον Αυτά τα ζητήματα θα είναι επίμαχα των οδικών δικτύων ε, σε σχέση με τις συνδυασμένες μεταφορές πρέπει να ε, συγκριθούν. Ε, υπάρχει επίσης για παράδειγμα τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πρώτα πρώτα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και την εισηγήτρια για την πρωτοβουλία αυτής της έκθεσης συμφωνούμε με τους τακτοποίηση τέλο πάντων του κλάδου και για τα κίνητρα ε, επίσης συμφωνούμε πέραν τώρα αυτών συμφωνούμε ότι θα πρέπει να γίνει μεταρρύθμιση να αλλάξει η ρύθμιση να αλλά ακόμα και η φρασιολογία γιατί από το 92 πράσαν πολλά χρόνια θα δείχνει δηλαδή πως γιατί μέχρι τώρα δεν μπορέσαμε να έχουμε μία αποτύπωση του τοπίου. Δηλαδή να αποτυπώσουμε το πώς έχει το τοπίο, πώς έχει, να μην έχουν πια αυτές τις ζώνες της συμφόρησης. τα των μελών και να δούμε τι θα γίνει με την υποδομή και σε σχέση με αυτό το πρόβλημα. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει με το άρθρο 3 εκεί που λέει ποιες είναι οι προϋποθέσεις του να έχουμε εξαντλητικούς ενδελεχείς. Όποτε υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις ε, θα πρέπει να αφαιθεί αυτό στα κράτη-μέλη. Μα ποιες είναι αυτές. Όποτε υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις ε, θα πρέπει να αφαιθεί αυτό στα κράτη-μέλη. Μα ποιες είναι αυτές οι συνθήκες ο καθένας θα το ερμηνεύσει αλλιώς. Δεύτερον, στο άρθρο 5, στο άρθρο 5 λέει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συντονιστούν με τα όμορα κράτη-μέλη τους για να υπάρχει σωστή εφαρμογή, να υπάρχουν επαρκείς εγκαταστάσεις και η άλλη μια φορά εδώ αναφέρεται το βασικό δίκτυο. Πώς θα επιληθεί το πρόβλημα. Και τέλος Πρόεδρε, εκεί που λέγεται τις εθνικές αρχές αναφέρεται ότι θα μπορεί να είναι σε αρμόδιες πάνω από μία αρχές βάσει όλα τα στοιχεία να υπάρχει εναρμόνιση να υπάρχουν τα δεδομένα και ο Ευχαριστώ κυρία Μπιλπάο. Η κυρία Κίλωνεν από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Πρόεδρε. Χαίρομαι λοιπόν που βλέπω μία νέα γνωμοδότηση μεταφορών. Θα ήταν καλό και για το περιβάλλον. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να διευκρινίσει πώς ε, βλέπει την χρηματοδότηση του τους με τα εφιστάμενα συστήματα μεταφορών. Για αυτά χρειάζεται να γίνει διάλογος. ώστε όλες οι κινήσεις να... Ευχαριστώ και εκ μέρους του Γιάκοπ Ταλούντε ε, για, ε, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά δεν βλέπω να λέτε γιατί δεν γίνεται. Εδώ και 20-30 χρόνια ζητούμε την μετακίνηση, τη μεταφόρτωση δηλαδή, από την οδική μεταφορά στο σιδηρόδρομο. Τα λεφτά είναι το πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει μαζικά στην κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, όπως και χωρισμένοι βεβαίως, και, δεν, και μένει απ' έξω ο σιδηρόδρομος τα τελευταία τρία χρόνια αυξήθηκαν τα διόδια στο σιδηρόδρομο 16% και όσο εξακολουθεί να υπάρχει αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός υπέρ των οδικών μεταφορών όποιες εκθέσεις και να γράψετε δεν περνώντας από την Αυστρία διότι είναι φθηνότερα. Το, προ... το παράδειγμα της Κλάουδια Σμίτη με τις Ηνωμένες Πολιτείες το ίδιο είναι έχουν ένα συνδυασμένο σύστημα 50% χωρίς πολύ. Υποστηρίζει χρηματοδοτικά την κατασκευή της τον σιδηρόδρομο ή από τον ε, πλωτό δρόμο θα αναπαυθεί ούτως ή άλλως ο, ο οδηγός. Υπάρχουν αυτά, αλλά δεν υποστηρίζεται επαρκώς. Να, εδώ θα ήταν μια σημαντική πρόοδος να το πετύχετε. Και εκεί όμως από τον αυτοκινητόδρομο επιβαρύνοντας και την οικονομία και το κλίμα και όλα. Ευχαριστώ κύριε Κράμερ. Κύριε Ντεμές Μάκερ. Κόσμο με ιδιαίτερα πυκνό κατοικημένη. Αλλά και ε, πραγματικά άξονα για τις ε, μεταφορές. 9% από 9% ε, του ΑΕΠ μας προέρχεται από την εφοδιαστική. Αυτή η πρόταση της Επιτροπής είναι σημαντική για μας. Χθε, μάλιστα, επισκέφθηκα έναν εμπορευματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στο κανάλι Αλμπέρ, εδώ στο Βέλγιο, και το οποίο έχει καλές κριτικές. Κάνει καλά πράγματα, αλλά έχει ακόμα πολύ μεγάλο δυναμικό. Ίσως μάλιστα και ανεπιθύμητο, όταν από τη μια μεριά υπάρχουν οι γενικοί κανόνες για το καμποτάζ και αυτοί γίνονται πιο αυστηροί, από την άλλη μεριά στην παρούσα οδηγία πηγαίνετε να ανοίξετε πάλι ένα παραθυράκι. Αυτό προκαλεί σύγχυση και ενισχύει τις καταχρήσει. Λέτε και το συνδυασμό με τις οδικέ μεταφορές. Γιατί δεν προωθείτε τις μεταφορτώσει στι πλωτέ σιδηρόδρομο, που είναι προφανής η στον σιδηροδρομο που ειναι προφανή ωφελεια Κατά τα λοιπά, οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέσεως της κυρίας Αγιούτο, θα έχει εκεί την ευκαιρία να παρουσιάσει την εκθεσή της και να τη σχολιάσει. Προθεσμία καταθέσεως τρόπο για προκαταρκτική ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον εισηγητή και τους και για προκαταρκτική ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον εισηγητή και τους και για την θέσπιση κοινών κανόνων για την πρόσβαση στην αγορά μεταφορών με λεωφορεία Πούλμαν. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, καμποτάζ, διασυνδέσεων κλπ. Η πρόθεση εδώ είναι να ολοκληρωθεί η αγορά μεταφορών με λεωφορεία ως εναλλακτική λύση στις μεταφορές με ιδιωτικά αυτοκίνητα. Πρώτα λοιπόν θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία προσωπεί εδώ ο κύριος Λιεζουά. Σας ευχαριστώ. Μπορείτε να λάβετε το λόγο για να παρουσιάσετε με λίγα, σε λίγα λεπτά την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2017 σε σχέση με τις υπηρεσίες πούλμαν ε, και λεωφορείων ε, Ξέρετε, ο ΜΑΝ σε μεγάλες αποστάσεις σε όλη την Ευρώπη θα, θα δώσει μια εναλλακτική επιλογή στη χρήση των ιδιωτικών οχημάτων και ελπίζουμε ότι θα συνεισφέρει στη μη φορείς, ε, σύλλογοι, συνδικάτα είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και τις απόψεις τους σε σχέση με την πρόταση αυτή. Επίσης έγινε και αξιολόγηση αντικτύπου και μελέτη ε, βάσει των οποίων ε, προέκυψε η πρόταση αυτή. Όπως είπα λοιπόν στόχος της πρότασης είναι να διευκολύνει την παροχή εμπορικών ε, τέτοιου είδους μεταφορών μεταξύ των της εταιρείες λεωφορείων από το να αναπτύξουν ε, νέες εμπορικές υπηρεσίες ε, μεταξύ των άστεων και επίσης το θέμα των τερματικών σταθμών και των, της διακριτικής μεταχείρισης που δεν δίνει τη δυνατότητα στους φορείς εκμετάλλευσης των λεωφορείων και οι σχετικές πρακτικές υπάρχει ένα ε, μια, ε, μια ε, ένα με ένα παζλ, ας πούμε, ένα ψηφιδωτό διαφόρων κανόνων που σημαίνει ότι είναι πάρα και γι' αυτό ακριβώς το πακέτο λέει ότι υπάρχει ανάγκη κοινών κανόνων. Κάτι ακόμη το οποίο είναι πολύ ευαίσθητο είναι η σχέση μεταξύ των εμπορικών υπηρεσιών και του των δημοσίων υπηρεσιών. Ε, Βεβαίω ε, θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ώστε οι εμπορικέ υπηρεσίε υπηρεσίας υπηρεσία που παρέχεται βάσει δημοσίων ε, δαπανών και επίσης τα κράτη-μέλη πρέπει να διατηρήσουν ε, ε τη δυνατότητα να ορίσουν τις υπηρεσίες που θα έπρεπε να καλύπτονται από την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας και τα κράτη αδειοδότησης και τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν αυτήν την αδειοδότηση αν θεωρούν ότι οι εμπορικές υπηρεσίες μπορούν να διακυβεύσουν την οικονομική βιωσιμότητα της ε, ε, υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας και ε, της υπηρεσίας της ίδιας. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε σαφείς κανόνες, αλλά είναι σημαντικό να υπάρχει και η απαραίτητη επιβολή της νομοθεσίας. Γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας εθνικός επόπτης που να εξασφαλίζει ότι οι κανόνες εφαρμόζονται ε, σωστά και αυτός ο έλεγχος να γίνεται με ανεξάρτητο τρόπο. Αυτή η απέτηση λοιπόν εθνικής εποπτείας ε, δεν θα οδηγεί σε διοικητικό κόστος για το κράτος μέλος. Ξέρετε ότι υπάρχουν ήδη επόπτες ε, μεταφορές. Συγγνώμη. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Έχουμε, μία, έχουμε μπροστά μας ένα έγγραφο το οποίο θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε επαναστατικό Πρόκειται για μια εξέλιξη πάντως των ε, υφισταμένων κανόνων αγορές τους, ε, με τελευταίες ε, πιο πρόσφατα τη Γαλλία και τη Γερμανία. Θα θέλαμε λοιπόν αυτή η πρόταση να συνεχίσει να πιέζει προς τη γενίκευση αυτής της τάσης και ελπίζουμε ότι η διαδικασία αυτή θα λάβει χώρα βάσει κοινών σαφών κανόνων για όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο εισηγητή μα τώρα θα λάβει το λόγο. Ο κύριο Ζήλε Ρομπέρ έχει εκείνο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εκπρόσωπο τη DigiMove. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε στο μέλλον κατά αυτόν τον τρόπο. Εγώ είμαι υπέρμαχο τη ε, ενιαία αγορά. Να σα υπενθυμίσω όμω ότι οι υπηρεσίε ε, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, τμήμα του ΑΕΠ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα πολύ σημαντικό τμήμα των μεταφορών, το, ένα πολύ σημαντικό τμήμα είναι και οι οδηγέ μεταφορέ. Υπάρχουν κάποιοι ε, ε, τομείς οι οποίοι καθυστερούν σε σχέση με την ολοκλήρωση τη ενιαία ε, αγοράς. Είναι μια φθηνότερη λύση η οποία δεν θα είναι όμως ει βάρο της ποιότητα της υπηρεσία. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μια υποφελή λύση για όλου σε άλλη χώρα από, την, ε, χώρα, από το σημείο το οποίο ξεκινάει ε, και δεν πρέπει να είναι αντικείμενο σε αυτή η περίπτωση. Δεν μπορούν ε, επόπτες, σε κάποιες χώρες ήδη υπάρχει υπάρχουν τέτοιου είδους ανεξάρτητες αρχές, σε άλλες χώρες δεν υπάρχουν. Πάντως να υπάρξει ένα τέτοιο σύστημα ακόμη και στο σιδηροδρομικό τομέα. Ε, εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Νικού φορέα, ε, μια διαδικασία επίλυσης. Τι μπορούμε να περιμένουμε. Κατά τη γνώμη μου θα υπάρξει πίεση κατά της ε, πρότασης αυτής από κρατημένες και πολλά, Κατά τη γνώμη μου, η βασική ανησυχία είναι η υποχρέωση παροχή δημόσια υπηρεσία. Θα αφορούν κυρίω τι μεγάλε αποστάσει. Κάθε κράτο μέλο ε, θα πρέπει να παρέχει περισσότερε επιδοτήσει από τα λεφτά των φορολογουμένων. Αυτό είναι πάρα πολύ επώδυνο ζήτημα. Πρέπει όμω να βρούμε ένα, μια λύση για να μην ε, ε, καταστρέψουμε την ουσία της πρότασης τη επιτροπή. Κάτι σε μερικά κράτη-μέλη ε, η σταθμή αυτή ε, ε, είναι αντικείμενο ε, αδειοδότησης από τους Δήμους, σε άλλες χώρες όχι, όπου μια εποφελή αγορά ε, μεγάλων διαδρομών ε, στον τομέα αυτό των οδικών μεταφορών. Υπάρχουν χώρες τις οποίες είναι πιο σε αυτές οι αγορές, σε άλλες χώρες λιγότερες. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα γενικότερο πλαίσιο, αν υπάρχει πίεση να υπάρξουν νέοι κανόνε για κάποια κράτη-μέλη, πρέπει να καταλάβουμε ότι για μερικού είδου υπηρεσίες, γιατί ακριβώ δεν θεωρείται πολύ κερδοφόρα αυτή η επιχείρηση. Συνοψίζοντας, θα ήθελα να σας πω ε, ότι ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συμβιβαστούμε, να βρούμε ένα συμβιβασμό για τα δύσκολα ζητήματα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μέχρι το κοινοβούλιο και θέλουμε να ακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ θα ακούσουμε τώρα τους και ηγητές για τρία λεπτά πάντοτε παρακαλώ. Παρακαλώ. Grandis Πασκουάλ του Λαϊκού Κόμματος. Grandis Πασκουάλ του Λαϊκού Κόμματος. Επανάσταση ή εξέλιξη είναι, ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπατε ότι είναι εξαίρεση, δεν το νομίζω την περασμένη εβδομάδα και μας είπε για την ουσία ποιο είναι το πρόβλημα. Ε, διατύπωσε διπλωματικά και πολύ διακριτικά. Η συγκεκριμένη πρόταση επομένω δεν έχει ε, αναλογικότητα. Έχει επικουρικότητα μόνο. Λέει εδώ πέρα για... Κοιτάξτε, το θέμα είναι να υπάρχει συμβίωση φυσιολογική μεταξύ διαφορετικών τρόπων μεταφοράς ο πιο κοινωνικός τρόπος. Ε, μπορούσε κανένας να πάει στα πιο μακρινά, στα πιο φτωχά, στα μη προνομιούχα μέρη. Ε, γι' αυτό και αυτό γίνεται πάρα πολύ συχνά με υποστήριξη οικονομική επιδότηση του κράτους ή με επιδότηση τέλο πάντων από άλλες πηγές. Η γωνία της χώρας. Το λεωφορείο θα πρέπει να συζητήσουμε πάρα πολύ το πόσο δίκαια είναι αυτά τα μέτρα, αυτέ οι προτάσεις. Ε, ανοιχτό διάλογο, είπε ο εισηγητή. Έτσι πρέπει να γίνει. Να κάτσουμε και να τα συζητήσουμε για αυτό το δύσκολο και σημαντικό θέμα. Η Επιτροπή Προπολογισμών είχε πολλές ε, επιφυλάξεις. Έχω και εγώ. Περίπλοκο το θέμα, δύσκολο. Οπότε όπου υπάρχει συναρμοδιότητα εθνική και κοινωτική για τις μεταφορές θα πρέπει να προσέξουμε να μην, ανατρέπουμε κάποια αποτελεσματικά συστήματα τα οποία εύρυθμα δουλεύουν. Ευχαριστούμε κύριε Ντεγκράντες Πασκουάλ. Κύριος Κουρομπάσεφ. Τον σωσικενή δεν γνωρίζω για ποιο λόγο, ίσως λόγω βουλγαρικής προεδρίας. Θα ήθελα βέβαια να μπορώ να μιλήσω στη γλώσσα μου. Αλλά θα κάνω μια παρατήρηση. Να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες της ε, φιλελευθερωποίησης και αν μας ικανοποιούν αυτές. Διότι αν ακολουθήσουμε για παράδειγμα το γερμανικό μοντέλο, ποιο είναι το αποτέλεσμα της απελευθέρωσης αυτής έχετε τελικώ εκεί μια εταιρεία η οποία κατέχει το 90% της αγοράς. Αν δηλαδή η απελευθέρωση οδηγήσει σε ένα σχεδόν μονοπόλιο, αυτό μας ενδιαφέρει να κάνουμε το ίδιο και στις άλλες χώρες μέλη. Ή αν έχουμε το καλό παράδειγμα της Ισπανίας, όπου υπάρχει συνδυασμό κερδοφόρων και μη κερδοφόρων γραμμών, είναι πολύ καλύτερα τότε να ανοίξουμε την αγορά, όταν ανοίξουμε την αγορά μάλλον, Χρειάζεται προσοχή να μην έρθει μια μεγάλη ε, αλλοδαπή εταιρεία και πάρει όλες τις κερδοφόρες γραμμές, όλες τις κερδοφόρες συνδέσεις και τελικώς φορτωθούν οι τοπικές κοινότητες και το κράτος την συντήρηση των μη κερδοφόρων γραμμών. Με την ίδια πρόταση απελευθερώνουμε και το καμποτάζ. Και εδώ πλέον έχω μπερδευτεί διότι στις εμπορευματικές μεταφορές θέλουμε να μειώσουμε το καμποτάζ, θέλουμε όμως να το απελευθερώσουμε στις ε, επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία. Είναι... Αυτή είναι η ερώτησή μου για το καμποτάζ και η ερώτηση για την απόσπαση των εργαζόμενων και τις διαφορές ανάμεσα σε επιβατικές και, εφορ... και ε, εμπορευματικές μεταφορές. Ασφαλώς και υπάρχει κίνδυνος εκεί. Το επόμενο είναι το όριο των 100 χιλιόμετρων απόσταση 100 χιλιόμετρων εδώ στο Βέλγιο, ε, στην ουσία σημαίνει διεθνείς μεταφορές. 100 χιλιόμετρα στην Ισπανία, στη Γαλλία δεν είναι καμιά σπουδαία απόσταση. Νομίζετε ότι όντω χρειαζόμαστε τέτοιο όριο και το όριο αυτό μπορεί να εφαρμόζεται σε κάθε χώρα μέλος ή θα αποδώσει σε κάθε χώρα μέλος με τον ίδιο τρόπο. Θεωρείτε ότι έχουμε κάποιες χώρες μέλη όπου είναι πολύ εξελιγμένη η αγορά των μεταφορών, τότε εκεί τις βοηθεί αυτής, αυτές η πρότασή σας. Εγώ δεν νομίζω. Μέλος όπως είστε εσείς θα πρέπει να το έχει δηλώσει εκ των προτέρων στην γραμματεία. για να δουν αν ίσως υπάρχει η ε, γλώσσα αυτή που έχει προβλεφθεί για τακτικό μέλος. Αυτό εξηγεί για ποιο λόγο είστε απογοητευμένος. Τώρα, δικές. τα προβλήματα που τέθηκαν το ίδιο δηλαδή πάντοτε ότι δεν θέλουμε ένα ιδιωτικό μονοπόλιο να υποκαταστήσει το κρατικό και για την δική μου ομάδα πάντως η αγορά, το άνοιγμα των αγορών είναι κάτι το ευκταίο και λόγω ελεύθερου ανταγωνισμού αλλά και για να ανοίξει και για να την σιδηροδρομική αρχή. Και διότι η διαχείριση, τώρα αυτή την ερώτηση θέλω να την κάνω εγώ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όταν ομιλείται για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος των ε, μεταφορών και μάλιστα πριν καν από την παρούσα πρόταση συχνά το άνοιγμα της δημόσιας το άνοιγμα μιας υπηρεσίας λεωφορείων, στο δρόμο δηλαδή, γίνεται στο σιδηρόδρομο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το τονίσει κανεί. Τώρα, για τους τερματικούς σταθμούς υπάρχει διπλό πρόβλημα. Το ένα που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της ελεύθερης πρόσβασης σε τερματικούς σταθμούς δηλαδή, υπάρχει όμως και ένα πρόβλημα έλλειψης επαρκούς αριθμού τερματικών σταθμών. Δεν υπάρχει δηλαδή επί κ. Κουρούμπασεφ για το καμποτάζ και για τους αποσπασμένου εργαζόμενους. Δηλαδή άλλο το καμποτάζ στον δρόμο, άλλο στον σιδηρόδρομο και το ίδιο του εργαζόμενους. Βλέπει κανεί ότι υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία παραμένουν ανοιχτά αναμένω που ίσως βέβαια να μην είναι ο τάβρος στο ιαλοπολείο αλλά πάντως είναι ένα θέμα το οποίο θα προκαλέσει έντονες συζητήσεις. Εγώ θα ήθελα πάντως να επιτευχθεί μια ισορροπημένη λύση που να λάβει υπόψη την δημόσια υπηρεσία και τις υποχρεώσεις που οφείλουν να τηρούν αδεσιών αυτών. Θα δώσω τον, λόγο στον κύριο Κράμερ τώρα Μιχαήλ, έχει το λόγο για τους πράσινους. Ευχαριστώ και εγώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον εισηγητή και βεβαίω το θέμα είναι δύσκολο διότι βέβαια οι διαφορές μεταξύ, δεν τίθεται δηλαδή το θέμα των διαφορών μεταξύ των ένας ε, οδηγός λεωφορείου. αν δεν έχει αναπαυθεί αρκετά αποτελεί κίνδυνο και για τους άλλους και για τους επιβάτε του. Και καλά, στο μεταξύ όμω έχουμε φτάσει σε ένα μονοπόλιο το οποίο καθορίζει όχι μόνο τις τιμές αλλά και τις αποστάσεις. Ειδικά εκεί όπου είναι αναγκαίο, ιδίω ε, οι εταιρείε μεταφοράς. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζω και το λεωφορείο φτηνό, το οποίο όμως ρηπαίνει πολύ περισσότερο. 100% προς όφελός τους τις υποδομές, αλλά τις υποδομές να τις πληρώνει ο φορολογούμενος όχι ο χρήστη. Αυτό δεν είναι δυνατέ που χρησιμοποιούν το ποδήλατο. 44 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο στην Ευρώπη. Εγώ αν θέλω ωστόσο, λέω λοιπόν προς όλους τους σιδηροδρόμους, αντί να κάθεστε να θρυνείτε, να δείτε ποια είναι η πραγματικότητα. Πέρσι, λέω λοιπόν προς όλους τους σιδηροδρόμους, αντί να κάθεστε να θρυνείτε, να δείτε ποια είναι η πραγματικότητα. πέρσι, πέρσι για τα δικαιώματα των επιβατών. Και να με συμπαθάτε που ξεπέρασα λίγο το χρόνο. Δηλαδή, Μάικλ, ε, προτιμούσες να πάρεις ε, το λεωφορείο και όχι το τρένο. Καινούριο αυτό και φοβερό νέο. Ε, να δώσω τώρα στους ε, σκιώδεις συζητητές το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον κύριο Ζήλε. Μα σε κάποιε χώρε όπω η Ισπανία, ακριβώ λόγω τη διαμόρφωση του εδάφου, λόγω τη κατανομή του πληθυσμού στο, στο, στον ύπεθρο που ε, είναι ασύμετρος, το δίκτυο των ε, λεωφορείων είναι ύψο, στον ύπεθρο που ε, είναι ασύμετρος το δίκτυο των ε, λεωφορείων είναι η πιο ε, έχουμε το δίκτυο των λεωφορείων το πιο, το, το πιο ευρύ, το πιο πυκνό στην Ευρώπη μα είναι και θέμα τελικά τη φορά που υπάρχουν λοιπόν κάποιοι διαγωνισμοί για την ανάθεση των δρομολογίων ε, πάντα τα πράγματα πάνε καλά, είναι δίκαια. Και οι εθνικές αρχές, όπως και σε μικρότερο βαθμό οι περιφερειακές αρχές, είναι σημαντικό αυτό το θέμα και για το έλλειμμα. Άρα περισσότερο από το αυτοκίνητό μας τα λεωφορεία. Λόγω ποιότητας, τιμής κλπ και οι σχετικές παραχωρήσεις, όπως είπε ο κύριος Ζήλε, όπως είπε η Κομισιόν, θα πρέπει να γίνονται μέσω διαγωνισμών. Ε, αυτά που λέει η Κομισιόν